Σας καλωσορίζω όλους. Έχουμε μια μέσα διάταξη ε, έτσι αρκετά απλή σήμερα. Σας ζητώ να την εγκρίνετε και να ολοκληρώσουμε παρακαλώ ένα τέταρτο πριν τις 12 έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι να φτάσουμε έγκαιρα στην Ολομέλεια για να ψηφίσουμε. Αυτό σημαίνει ότι θα ολοκληρώσουμε στις 11.45. Την 3η 29 Μαΐου στη συνεδρίαση στο Στρασβούργο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τέσσερις νομοθετικές προτάσεις που αποτελούν τη βάση της νέας γενιάς της πολιτικής συνοχής μετά το 2020. Αυτές τις τέσσερις προτάσεις, όπως γνωρίζετε, αφορούν έναν κανονισμό με κοινέ διατάξεις ό,τι αφορά τα διάφορα ταμεία, το CPR, έναν κανονισμό που αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής, ένας κανονισμός για την ε, εδαφική συνοχή, το Interreg μετά το 2020 και ένα κανονισμό που προβλέπει ένα νέο μηχανισμό για τα διασυνοριακά project. Άλλες νομοθετικές προτάσεις όπως αυτές που δημιουργούν ε, το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα εγκριθούν αυτή την εβδομάδα και θα ακολουθήσουν και άλλες τις επόμενες εβδομάδες όπως η νέα εκδοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις στρατηγικές επενδύσεις και το πρόγραμμα στήριξης για την διαθροτική μεταρρύθμιση. Δεν έχουμε ακόμα λοιπόν μια πλήρη συνολική εικόνα όλων αυτών των εργαλείων που θα ε, διαμορφώσουν τη νέα πολιτική συνοχή της Ένωσης, συνοχής της Ένωσης. Όμως ε, τα βασικά στοιχεία, οι βασικοί κανονισμοί έχουν ήδη δημοσιευθεί. Καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ με μεγάλη χαρά την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, την Κορίνα Κρετού, την οποία ευχαριστώ που είναι εδώ μαζί μας και που είναι υπεύθυνη για τις προτάσεις που εγκρίθηκαν την περασμένη Τρίτη. Αναμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία τα σχόλιά σας, τις πληροφορίες σας για την πρόταση αυτή η οποία ε, έχει ήδη ανακοινωθεί. Θα δώσω το λόγο πρώτα λοιπόν στην Επίτροπο για μια αρχική τοποθέτηση 15-20 λεπτών. Στη συνέχεια θα πάρουν το λόγο τα μέλη της Επιτροπής μας για να σχολιάσουν και βέβαια ως συνήθως θα δώσω πρώτο λόγο στον, στους συντονιστές και μετά στα λοιπά μέλη. Και όπως σας είπα θα ολοκληρώσουμε στις 12 παρατέταρτο. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Σε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής θα σας εξηγήσω ε, το αποτέλεσμα μιας μακράς δύσκολης έντονης διαδρομής ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω ότι έχει υποβάλει μια ισορροπημένη πρόταση και για το επόμενο πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά και για την πολιτική συνοχής. Η πολιτική μας παραμένει ισχυρή για όλες τις περιοχές, για όλες τις περιφέρειες. Χρειάστηκε αποφασιστικότητα ε, όλων όσων προσπίζονται αυτή την πολιτική για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα αυτό. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την Επιτροπή Ρέτζι που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή και έδωσε μάχες για την πολιτική συνοχή. Δεν ήταν εύκολο. Όπως μόλις είπα, το νέο νομοθετικό πακέτο για την πολιτική συνοχή είναι ισορροπημένο, κατά τη γνώμη μου, στα πλαίσια βέβαια του Brexit και των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, πιστεύω ότι αποτελεί επίτευγμα Γνωρίσαμε τι περιμέναμε όταν δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή για το νέο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε ένα νέο ε, προπολογισμό φιλόδοξο 1,1 τρισεκατομμύρια ευρώ και στα πλαίσια αυτά η πολιτική συνοχής ε, παραμένει ε, μια σημαντική πολιτική επενδύσεων είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Ευθύ εξ εγώ θέλησα να εξασφαλίσω ότι οι πόροι της πολιτικής συνοχής θα κατανεμηθούν αναπεριφέρεια και αναχώρα όσο γίνεται πιο δίκαια. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα προπολογισμό που επικεντρώνεται ε, σε αυτούς που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Επικεντρωνόμαστε περισσότερο από ποτέ ε, στις πιο φτωχές περιφέρειες των κρατών μελών αλλά και στις περιφέρειες με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, στις περιφέρειες που έχουν πληγεί περισσότερο από την, την προσφυγική κρίση και αυτούς που πλήττονται επίσης από ε, τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Όπως γνωρίζετε η πρότασή μας επίσης αντικατοπτρίζει την ε, υπόσχεσή μας να επικεντρωθούμε στις επενδύσεις μας εκεί όπου πιάνουν τόπο μια πιο εστιασμένη πολιτική συνοχής γενικότερα θα δείτε ότι έχουμε λιγότερους στόχους και πιο σύγχρονους. Λέω σύγχρονους διότι έχουμε δώσει εδώ έμφαση ε, σε ζητήματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ε, της ε, παγκοσμιοποίησης. Βιομηχανική ε, βιομηχανικός εξυγχρονισμός, περιβαλλοντικά φιλικές πολιτικές κλπ. Θέλουμε οι χώρε, οι περιφέρειε να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία για να επιλέγουν τι κατάλληλε επενδύσει. Επιπλέον έχουμε ε, ευρύτερου και λιγότερους στόχους, ε, μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών, μεγαλύτερη ευελιξία σε επίπεδο προγραμμάτων. Η ευελιξία έχει αυξηθεί και με τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση το 2025 όπου και θα μπορέσουμε να δούμε εάν θα πρέπει να αλλάξει κάτι για τα τελευταία δύο έτη. Αυτό βοηθάει την προσαρμογή διότι η εμπειρία μας μας έδειξε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα είναι τα πράγματα σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια ή πριν από 7 χρόνια δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε ότι θα λάβουν χώρα τόσες αλλαγές στην Ήπειρό μα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο ευέλικτοι στο πρόγραμμά μα. Ταυτόχρονα όμω θα πρέπει να είναι πιο γρήγορη η εφαρμογή. Γι' αυτό προτείνουμε να επανέλθουμε στον κανόνα νη συν 2 αυτό θα επιταχύνει την εφαρμογή έτσι ώστε οι πολίτες να δουν τις αλλαγές αυτές ε, με απτό τρόπο επιτόπου. Θέλουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά στον πολίτη και αυτό αποτυπώνεται και στο θεματικό μενού μας. Προτείνουμε μια, κάποιους πολιτικούς στόχους ε, που έχουν να κάνουν με την εδαφική διάσταση της συνοχής και κατά αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ε, την βιώσιμη αστική ανάπτυξη ε, και να δώσουμε γενικότερα περισσότερε εξουσίε στο τοπικό επίπεδο. Θέλουμε να έχουμε και μια πιο συνεχτική προσέγγιση ό,τι φορά τι πόλει. Υπάρχουν πολλά ε, εργαλεία ε, αστικού τύπου για τι πόλει δηλαδή. Υπάρχει αυτή η ατζέντα. Αλλά είναι κατακαιρματισμένα αυτά τα εργαλεία και ορισμένε φορέ είναι δύσκολο οι τοπικέ αρχέ να γνωρίζουν πού θα βρουν στήριξη. Προτείνουμε λοιπόν ένα ενιαίο πλαίσιο, την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία με διάφορα εργαλεία, το Urban ε, και αυτό και το δίκτυο ε, ανάπτυξη Urban, το αστικό. Από το... Στο μέλλον λοιπόν θα μπορούν τα, οι πόλεις να έχουν λόγο στο πώς ε, αναπτύσσονται να μην εξαρτώνται από τις Βρυξέλλες ή από το Λουξεμβούργο, διότι αυτοί γνωρίζουν καλύτερα. Αυτή η εδαφική διάσταση αποτυπώνεται και μέσω της ε, διαπεριφερειακής συνεργασίας. Είναι η πιο απτή έκφραση του ευρωπαϊκού αυτού σχεδίου και εκεί είμαστε φιλόδοξοι. Πρώτα απ' όλα προτείνουμε η διαπεριφερειακή συνεργασία να είναι οριζόντια προτεραιότητα, θα αφορά δηλαδή όλους τους πολιτικούς στόχους, όλους τους στόχους πολιτική και γι' αυτό λοιπόν η συνεργασία ε, πέρα από το κάθε πρόγραμμα θα είναι πιο απλή. Επίσης υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία όπως ε, καινοτόμε επενδύσεις διαπεριφερειακά ε, για να βοηθήσουμε ε, τις περιοχές που θέλουν να εξειδικευθούν με έξυπνο τρόπο. Θέλουμε επίσης να μπορέσουμε να προσπεράσουμε τα διοικητικά, τα γραφειοκρατικά εμπόδια σε διασυνοριακό επίπεδο, να είναι πιο απλά τα διασυνοριακά project, έτσι ώστε εθελοντικά ε, να μπορούν να ακολουθούνται οι κανόνες ενός κράτους μέλους και σε ένα άλλο γειτονικό ελπίζουμε αυτό να διευκολύνει τα πράγματα κατά την εφαρμογή των διασυνοριακών προγραμμάτων συνεργασίας εφόσον βέβαια ένα κράτος μέλος ε, δεχθεί την νομοθεσία του άλλου ε, βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η πρόταση μας επιτρέπει να είμαστε φιλόδοξοι αλλά και ρεαλιστές αν θέλουμε οι επενδύσεις στον τομέα της συνοχής να κάνουν τη διαφορά, χρειαζόμαστε απλούς τρόπους εφαρμογής τους. Αυτό το νέο νομοθετικό πακέτο θα μας οδηγήσει εκεί κατά τη γνώμη μου και μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω ότι έχουμε εργαστεί σκληρά επ' αυτού. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ βεβαίω και τις υπηρεσίες μου. Ε, οι προϋποθέσεις για τις επενδύσεις τώρα, εδώ έχουμε τις προϋποθέσεις ex ante και υπάρχουν αυτές τις προϋποθέσεις ε, που δημιουργούν τη δυνατότητα έχει μειωθεί κατά το ίμιση. Ε, ο, ο κατάλογος, είναι, τα κριτήρια είναι πολύ πιο απτά. Υπάρχει ένας κατάλογος επίσης μέτρων απλοποίησης όπως ε, το τέλος ε, της διαδικασίας ορισμού απλουστευμένες επιλογές ότι αφορά το κόστος, επέδο ελέγχου βεβαίως θα πρέπει να ελέγχουμε το πόσο ε, χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα των φορολογουμένων, απλοποιημένε διαδικασίε και εδώ για τα προγράμματα τα οποία έχουν καλό ποινικό μητρό, αν θέλετε, λευκό ποινικό μητρό. Ε, θα γίνουν, θα γίνουν επίσης και αναλύσει αξιολογήσεις κινδύνου και να έχουμε, για να έχουμε ενιαίους ελέγχους. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα επίπεδα ελέγχου. Υπάρχει το ελεγκτικό συνέδριο, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να το αποφύγουμε αυτό Θέλουμε να επικεντρωθούμε κυρίως στο έργο των υπάρχοντων οργάνων, έτσι ώστε ο τελικός να μην ε, επιβαρύνεται από τους πολλούς ελέγχους. Δεν θέλουμε απλά να συλλέγουμε ε, κάποιους λογαριασμούς, δεν θέλουμε μόνο διαδικασίες, δεν θέλουμε διοικητική επιβάρυνση, θέλουμε ε, αποτελέσματα, θέλουμε την οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Θέλουμε πιο απλά συστήματα χρηματοδότηση. Για πρώτη φορά ευθυγραμμίζουμε ε, τα οικονομικά μέσα και τις ε, ενισχύσεις έχουμε κοινούς κανόνες ε, που είναι μισή από αυτούς που υπάρχουν τώρα η όλη δομή είναι πιο συνεκτική προτείνουμε κοινέ διατάξεις για κοινή διαχείριση κάποιων ταμείων αυτό θα οδηγήσει σε μια πιο συνεπή προσέγγιση ό,τι αφορά την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση Ελπίζω αυτό να μειώσει το διοικητικό άχθος για τις αρχές αλλά και τους δικαιούχους. Επίσης ε, έχουμε θεσπίσει νέους τρόπους ε, για να μπορούμε να συνεισφέρουμε σε άλλα ε, ευρωπαϊκά μέσα όπως ορίζοντας 2020 το Εράσμους και το Invest EU. Αξιότιμα μέλη, αυτά είναι τα κύρια σημεία του νέου νομοθετικού πακέτου για την πολιτική συνοχή. Έχουμε ξεκινήσει μια φιλόδοξη διαδρομή απλοποίησης, ευελιξίας με βάση τις εμπειρίες του παρελθόντος ε, με βάση τα λάθη μας ε, χωρίς όμως να αλλάζει ουσιαστικά η αρχιτεκτονική ε, του συστήματός μας. ελπίζω να έχουμε ένα υποδομητικό διάλογο στις διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να ξεκινήσουμε έγκαιρα την νέα προγραμματική περίοδο. Σας διαβεβαιώ ότι ο πρόεδρος Γιούγκερ και εμείς ε, θέλουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαπραγμάτευση πριν τις Ευρωεκλογές, όχι λόγω των ευρωεκλογών βέβαια, αλλά διότι είναι ανάγκη να ξεκινήσει η εφαρμογή την 1η Ιουλίου του 2021 ε, ε, για να μην έχουμε τις καθυστερήσεις που είχαμε τώρα από τις μελέτες μας προκύπτει ότι αν δεν ξεκινήσουμε την 1η Ιουλίου 2021 την εφαρμογή πάνω από 150.000 προγράμματα ε, κινδυνεύουν να μην ολοκληρωθούν. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για το έργο σας, για την υποστήριξή σας, ε, την εμπιστοσύνη σας. Αναμένω να ακούσω τις απόψεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ας ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Θα δοθεί χρόνος ομιλίας στους συντονιστές και ξεκινάμε με το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να σας ζητήσω την άδεια ε, να μοιραστούμε το χρόνο ομιλίας με τον Γιάννη Ούλμπριχτ. Οπότε θα κάνω εγώ μόνο κάποιες προκατακτικές παρατηρήσεις. Σας ευχαριστούμε κυρία Επιτροπή που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Κρατήσατε την υπόσχεσή σας ότι θα επιστρέψετε με όλα τα θέματα για να μας δώσετε τη δυνατότητα να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Και σήμερα το πρωί στη συνάντηση των συντονιστών συμφωνήσαμε να ορίσουμε όλους τους εισηγητές τον Ιούνιο. όπως το κάναμε και για τον κανονισμό των γενικών διατάξεων, να ορίσουμε τους ε, συντονιστές τους ε, εισηγητές, συγγνώμη, για να αρχίσουμε τις εργασίες μας και να ολοκληρώσουμε την πρώτη εξέταση κατά την αρχική περίοδο. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν, έχουμε κάνει όλες τις προετοιμασίες. Έχουμε τις 7 εκθέσεις για τη συνοχή και υπάρχουν πολλά που μπορούμε να συζητήσουμε σε σχέση με όλα αυτά που μας παρουσιάσατε. Αλλά έχουμε κατά νου ε, και τα αποτελέσματα, ε, αυτά τα οποία θα πρέπει να ε, συναγάγουμε ως συμπεράσματα. Δεν μας είπατε πολλά για οικονομικά στοιχεία και θα δώσω το λόγο στο Γιάνν Όλμπριχτ. Ευχαριστώ. Είμαι η για το MFF, για την, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, και θα ήθελα να κάνω κάποιες, κάποιες σχετικές παρατηρήσεις. Το σύστημα υλοποίηση θα το συζητάει η Επιτροπή μα ε, κατά του επόμενου μήνε και είναι πολύ σημαντικό να βρούμε ένα καινούριο σύστημα. Αλλά δεν ξέρω ευτυχώ ή ατυχώ, άλλαξε τη διαδικασία η Επιτροπή. μιλούσαμε για μείον 7% για τη συνοχή χρησιμοποιώντα τα στοιχεία του 2020 σε τρέχουσε τιμέ, αλλά μετά ακούσαμε ότι η συνοχή θα μειωθεί κατά 10% σε τιμέ 2018. Αν είναι μείον 10% περιμένουμε στοιχεία. Ποιες είναι οι συνέπειες του μείον 10%. Μετά μας δόθηκαν στοιχεία μείον 46% για το Ταμείο Συνοχής και αυτό δεν είναι μικρή μείωση αν από το μείον 10 κόψουμε το Ταμείο Συνοχής κατά 46%, τα άλλα ταμεία θα αυξηθούν αναλογικά. Περιμένουμε λοιπόν να μας δώσετε και κάποια αριθμητικά στοιχεία. Πριν από δύο μέρες μας δώσατε κάποια στοιχεία ως παράρτημα για το κανονισμό κοινών διατάξεων που μας έκανε εντύπωση γιατί αυτό θα ψηφιστεί κατά πλειοψηφία. Τέλος πάντων έχουμε τα στοιχεία για τα εθνικά κονδύλια. Αρχίσαμε να αναλύουμε τα στοιχεία που μας δώσατε πριν από δύο μέρες και ανακαλύψαμε στοιχεία που μας εκπλήσουν. Μείον 24, μείον 23 κλπ. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν ποια είναι η μεθοδολογία. Πώς καταλήξατε σε αυτά τα νούμερα. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις. Και τώρα έχω και τις εξής ερωτήσεις. Πρώτον, σύμφωνα με την ανάλυση και τα στοιχεία που έχετε, ποιες είναι οι χώρες συνοχής σήμερα. Είναι οι ίδιες χώρες συνοχής ή θα έχουμε λιγότερες χώρες συνοχής στο μέλλον θα αλλάξει καθεστώς κάποια από τις χώρες και θα βγει από το Ταμείο Συνοχής. Αυτό θα εξηγούσε εν μέρη το μείον 46%. Δεύτερον, ο ορισμός των λιγότερων ενεπτυγμένων περιοχών. Ποιος είναι. Γιατί χρησιμοποίησατε το 80% του ΑΕΠ και 20% λοιπόν στοιχείων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Άρα, ο ορισμός των λιγότερων ενεπτυγμένων χωρών άλλαξε. Ο ορισμός της μεταβατικής ε, περίοδου επίσης έχει αλλάξει. Πέρασε από το 75% στο 90% του ΕΠ και μετά στο 100%. Δηλαδή κομμάτι των κάτω χωρών ε, γίνεται μεταβατικό. Το μεγαλύτερο κομμάτι της Γαλλίας επίσης είναι σε μεταβατική περίοδο. Το ποσοστό λοιπόν των λιγότερων επιτυγμένων προς τις χώρες σε μετάβαση έχει αλλάξει εντελώς. Σήμερα έχουμε ένα συγκεκριμένο ρυθμό λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών στην Ευρώπη. Στο μέλλον θα έχουμε τον ίδιο ρυθμό των λιγότερων ανεπτυγμένων περιοχών ή έχει αλλάξει το ποσοστό. Γιατί αν λέτε ότι η πολιτική συνοχή θα αφορά κυρίω τι λιγότερο ανεπτυγμένε, τι εννοείτε. Τι εννοείτε όταν λέτε λιγότερο ανεπτυγμένε περιοχέ. Καταλαβαίνουμε ότι αν σήμερα μιλάμε για 330 δισεκατομμύρια για την πολιτική συνοχής, τα στοιχεία της Επιτροπής χρησιμοποιώ. Αυτό δεν είναι για το κεφάλαιο της συνοχής, είναι η παραδοσιακή πολιτική. 330 δισεκατομμύρια για παραδοσιακή ε, πολιτική συνοχής. Ο τρόπος ε, κατανομής των 330 δισεκατομμύριων είναι, καταλαβαίνω εγώ, ότι θα είναι για τις λιγότερα ανεπτυγμένες ε, σε μετάβαση και γι' αυτό επαναλαμβάνω την ερώτησή μου. Ποιε είναι οι χώρε συνοχή, για να καταλάβουμε τι είναι το Ταμείο Συνοχή, τι έχει γίνει στο Ταμείο Συνοχή. Δεύτερη ερώτηση. Οι λιγότερο αναπτυγμένε περιοχέ έναντι περιοχών σε μετάβαση και των περισσότερων αναπτυγμένων περιοχών. Το 20% των επιπλέον κριτηρίων άλλαξαν εντελώ την κατάσταση. Και μία παρατήρηση. Φαίνεται να έχει αλλάξει η πολιτική όχι η υλοποίηση. Η πολιτική φαίνεται να έχει αλλάξει. Οι κατευθύνσει της πολιτικής φαίνεται να έχουν αλλάξει. Όντως υπάρχει τέτοια αλλαγή. Ή είναι η πολιτική εξόδου που δικαιολογεί τις μειώσεις αυτές. Ευχαριστούμε. Κωνσταντς Κρέλ, εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση που μας κάνετε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι θετικό. Χαίρομαι που και στο μέλλον η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι θα μπορούν να συμμετέχουν όλες οι περιφέρειες στην πολιτική συνοχή. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ήμασταν πάντοτε σίγουροι ότι θα μπορούσε να ισχύει αυτό. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό το σήμα το οποίο λαμβάνουμε από την Επιτροπή και ως Κοινοβούλιο μπορούμε να το μεταφέρουμε στους πολίτες της Ευρώπης. Θεωρώ πολύ θετικό ότι υπάρχει σαφώς υψηλότερη ευελιξία για τις περιφέρειες όσον αφορά τις προτεραιότητες οι περιφέρειες θα έχουν μεγαλύτερο δικαίωμα συμμετοχής για να μπορούν να δηλώσουν τις προτεραιότητές τους, ε, αυτά τα οποία ε, θεωρούν ζητήματα που θέλουν να επιλύσουν στην περιφέρειά τους. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό Ξεκινήσαμε με τον κανονισμό Omnibus για την ε, απλούστευση της πολιτικής, για λιγότερη γραφειοκρατία της πολιτικής συνοχής και ε, χαίρομαι που η Επιτροπή συνεχίζει σε αυτό το ρυθμό. Είναι σημαντικά μηνύματα και χαίρομαι και εγώ προσωπικά γιατί εγώ προέρχομαι από αστικό χώρο και θα μπορούν και οι ίδιες οι πόλεις να έχουν ισχυρότερο ρόλο και θα έχουν τη δυνατότητα να συμπροσδιορίζουν τις προτεραιότητες ε, σε σχέση με το παρελθόν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την πολιτική συνοχή κατά με είναι η μείωση, η σαφής μείωση του προϋπολογισμού και με ενοχλεί ότι ο κύριος Έρτιγκερ, αυτό δεν έχει σχέση με εσάς κυρία Κρέτσου, αλλά ο κύριος Έρτιγκερ δηλώνει ε, που υπάρχουν προβλήματα και για την πολιτική συνοχή καταλήγουμε να έχουμε λιγότερα χρήματα και υπάρχουν και περιοχές σε μετάβαση στις κάτω χώρες που είπε και ο Γιάννης που χάνουν ε, 22-23% των διορθωτικών ταμείων. Είναι δραστικές μειώσεις για ορισμένα κράτη-μέλη αυτές. Και χθε στο ψήφισμα για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο το Κοινοβούλιο κατέστησε σαφές ότι εμείς δεν συμφωνούμε με τέτοιες περικοπές. Και θα συνεχίσουμε να το διαπραγματευόμαστε αυτό το θέμα. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να δούμε και για το περιεχόμενο της πολιτικής συνοχής. Έχω δύο ερωτήσεις. Η ομάδα μου, αλλά και εγώ προσωπικά, δεν κατανοούμε γιατί η μακροοικονομική ερεσιμότητα είναι και πάλι κομμάτι του κανονισμού ε, ε, κοινών διατάξεων Εντάξει, έτσι και θα μπορούσαν και οι Ιταλοί συνάδελφοι να ρωτήσουν ε, κατά πόσο επηρεάζεται το κονδύλι και για την Ιταλία με βάση τον κανονισμό για τις ειδικέ διατάξεις. Θέλω να πω ότι δεν είναι το νόημα της πολιτικής συνοχής αυτό και από τα, τις εμπειρίες του παρελθόντος. Ξέρω ότι για την Ελλάδα είχαμε ένα ειδικό πρόγραμμα για να μπορεί να επενδύει με τα διορθωτικά ταμεία για να μπορέσει να βγει από την ε, κρίση. Προσπάθειες για την Ισπανία και την Πορτογαλία κάτω ε, ε, απέτυχαν αυτές οι προσπάθειες να τις βάλουμε κάτω από τον κανονισμό των ειδικών διατάξεων και τώρα φαίνεται σαν να το ξαναφέρνουμε ε, στο προσκήνιο. Και μια δεύτερη ερώτηση. Ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο έχει κάποιες επιφυλάξεις να γίνονται διαθωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη μέσω του Ταμείου Συνοχής. Μπορεί σημειακά να υπάρχουν κάποιες σχέσεις, αλλά δεν ισχύει στην πράξη αυτό. Η πολιτική συνοχή έχει διαφορετικά καθήκοντα και όχι τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Δεν ξέρω γιατί το ξαναφέρνουμε ως τμήμα της πολιτικής συνοχής. Και τρίτον, και αυτό αφορά και την παρατήρηση του Γιάνν, χαιρόμαστε να έχουμε διαφάνεια για τα εθνικά κονδύλια, τους εθνικούς φακέλους ε, στο παράρτημα για τον κανονισμό των ειδικών διατάξεων, διευρυμένη μέθοδος του Βερολίνου, αλλά είναι πρώτη φορά που αυτό γίνεται στο πλαίσιο του κανονισμού ειδικών ε, ε, κοινών διατάξεων. Δεν ξέρω αν είναι δικό μας καθήκον να εξετάζουμε το αν θα πάρουμε κάποια ποσοστά παραπάνω για την πολιτική απασχόληση, για την ενεργεία των νέων, για την απασχόληση των γυναικών, για τους πρόσφυγες. Υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούμε σε αριθμητικά στοιχεία που διαπραγματεύονται οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και οι κυβερνήσεις. Δεν θέλουμε να τους βάλουμε το μαχαίρι στο λαιμό και να πούμε ότι πρέπει τώρα να αποφασίσετε στο Κοινοβούλιο για την κατανομή του προϋπολογισμού. Δεν είμαι βέβαιη ότι έχει νόημα να ακολουθήσουμε αυτή την τακτική. Και ε, μία ε, επιπλέον παρατήρηση. Ελπίζω ότι ε, για το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε σχέση με τον κανονισμό κοινών διατάξεων αυτό το οποίο προτείνεται να μην οδηγήσει σε προβλήματα για την Ήπεθρο και οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Γεωργίας θα πρέπει να έχουν κατά νου την προοπτική της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στο μέλλον. Ε, χάσαμε τα σχετικά με το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αν μπορείτε να κάνετε κάποιο σχετικό σχόλιο θα σας ήμουν ευγνώμων. Ευχαριστώ. Τόμασικ για την ECR. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε που είστε ξανά μαζί μας σήμερα. Σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει χώρες που δεν έχουν αποκτήσει αρκετή εμπειρία και τεχνογνωσία προκειμένου να υποβάλουν έτσι για τον ορίζοντα 2020 και για άλλα ταμεία της, από την κεντρική διοίκηση. Εξαιτίας του Brexit και της ε, έλλειψης επαρκών πόρων στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα ταμεία τα οποία χάνουν κεντρικής διαχείρισης. Οπότε η ερώτησή μου είναι η Κομισιόν θα βοηθήσει και πώς θα βοηθήσει τα πιο καινούρια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα την Κροατία η οποία εντάχθηκε το 2013 στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις. Πώς θα βοηθήσετε αυτές τις χώρες προκειμένου να μπορέσουν να απορροφήσουν περισσότερα, περισσότερους πόρους. Πολύ δε περισσότερο που το Ταμείο Συνοχής ε, θα δει να περικόπτονται οι πόροι του κατά περισσότερο από 45%. Merci. Pour le groupe euh, Ματίς Φαν Μίλτεμπορκ για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ μαζί μας δύο μόλις μέρες μετά την παρουσίαση των προτάσεών σας. Ε, μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από αυτό που βλέπω. Θα ενισχύσετε ε, την σύνδεση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Ξάμεινο και την πολιτική συνοχή. Πάντοτε το υποστηρίζαμε, συμπεριλαμβανομένων και των μακροοικονομικών αιρεσιμοτήτων που βελτιώνονται διότι πλέον λαμβάνεται υπόψη και την διαδικασία μακροοικονομιών ανισορροπιών. Οπότε αυτό θα βελτιώσει την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Το καλωσορίζουμε, παρόλο ότι μπορεί να είμαστε ε, ε, αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα πιστούν και οι υπόλοιποι, γιατί αυτό είναι αυτή είναι σωστή ε, κατεύθυνση. Μετά έχουμε τον ΙΣΙΝ 2 και την επιτάχυνση των διαδικασιών και αυτά καλά. Και έχουμε και την καινούργια δραστηριότητα Urban. πολύ καλό να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε με, την, ε, ε, με το θεματολόγιο Urban. Ε, μετά, προτείνονται ε, καινοτόμες επενδύσεις, διαπεριφερειακές επενδύσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για την Ευρώπη προκειμένου οι περιφέρειες μας να γίνουν ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί δεν μιλούμε μόνο για τη συνοχή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ιδέα λοιπόν της διεύρυνσης του Interreg Europe, του πεδίου εφαρμογή του, με την δυνατότητα να γίνονται επενδύσεις, πραγματικές επενδύσεις στην πραγματική οικονομία και να δημιουργούνται αλυσίδες αξίας. Έχω όμως και ορισμένες ερωτήσεις διότι έχουμε ζητήσει επανειλημμένως ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και το Κοινοβούλιο στο σύνολό του να αυξηθεί ο προπολογισμό του Interreg. Και με έκπληξη μου βλέπω ότι ε, ο φάκελος, ε, το ποσό για την ε, χωρική συνεργασία θα μειωθεί κατά 16,5% ίσως και περισσότερο, ξέρετε πώς θα το υπολογίσουμε στην, επιτροπή, στην έκθεση Ζουλό και στην έκθεση Βέστφαλ δεν είχαμε πει αυτό, είχαμε ζητήσει αύξηση. Καταλαβαίνω ότι θέλετε ε, ειδικά ο, χρηματοδοτικά εργαλεία ε, όπως αυτό το προενταξιακό να, το να τα βάλετε όλα στο ίδιο ε, ταμείο αλλά έχουμε και κάποιους στόχους του Interreg. Ένας από αυτούς τους στόχους είναι μια πιο ασφαλής Ευρώπη δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο βασικός λόγος για την εδαφική συνεργασία στην Ευρώπη είναι να ε, ξεπεραστούν τα σύνορα, ιδιαίτερα τα εσωτερικά σύνορα, αλλά και τα σύνορα με τρίτες χώρες. Ε, το θέμα δεν είναι η αστυνόμευση των εξωτερικών σύνορων, οπότε μπορείτε να μας διευκρινίσετε τι είδου ε, προγράμματα θα... Ε, χρηματοδοτηθούν, ε, ιδιαίτερα δεδομένου αυτού του καινούργιου στόχου Ιντερεκ περί ασφαλέστερης Ευρώπης. Δεν είμαι σίγουρο ότι πρέπει με ευρωπαϊκά χρήματα ε, να χρηματοδοτήσουμε και άλλους φράχτες στα εξωτερικά σύνορα. Η άλλη μου ερώτηση αφορά το απόθεμα επίδοση. Μετά από μια πρώτη εξέταση βλέπουμε ότι αυτό συνεχίζεται ε, στην επόμενη πραγματική περίοδο. Για ποιο λόγο, δεδομένου ότι δεν έχουμε και καλή εμπειρία. Έχουμε ακόμα το τρέχον έτος πριν καταφέρουμε να εξετάσουμε το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το απόθεμα επίδοση σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Οπότε λοιπόν ποια είναι η έννοια του να συνεχίσουμε ε, να το χρησιμοποιούμε ε, χωρίς να έχουμε την αξιολόγησή του. Μετά, ε, τους λογιστικούς ελέγχους και τις ε, επιβεβαιώσεις ε, διαχείρισης ε, των προγραμμάτων. Καταλαβαίνω τις βελτιώσεις προσπαθεί να φέρει η Κομισιόν σε αυτό το θέμα και να μειώσει τη γραφειοκρατία, αλλά θα ήθελα να μου πείτε πώς, τι θα γίνει στην πράξη. Ποιος θα αξιολογήσει το κατά πόσον μπορεί να ε, απλοποιηθεί για την Α ή τη περιφέρεια η απλοποίηση. Η Κομισιόν θα το αποφασίσει, θα εξαρτάται από το ποσό του προγράμματος που χορηγείται, από το συνολικό ποσό που λαμβάνει κάθε χώρα, από την εμπειρία που είχατε από την Α ή τη Β χώρα τα τελευταία χρόνια. Πώς θα δοθεί αυτή η διευκόλυνση. Γενικά λοιπόν συμφωνώ με κανοποιούν προτάσεις, εξυγχρονίζεται η πολιτική μας Πρόκειται για μια εξέλιξη, όχι μια επανάσταση, το είπα και παλιότερα και πολύ καλό αυτό, γιατί ε, αν ξεκινούσαμε μια επανάσταση δεν θα επιτρέπαμε σε όλες τι επιχειρήσεις, σε όλες τι περιφέρειες, σε όλους πολίτες να υποφεληθούν. Νομίζω ότι ο στόχος μας είναι μια Ευρώπη η οποία θα πρέπει να δίνει αποτελέσματα εμφανή και ορατά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ματής. Μονίκα Βένε για τους πράσινους. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και την Επίτροπο που είναι εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε την πρόταση που υποβάλλατε πριν από μερικές μέρες. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω με κάτι θετικό. Για άλλους λόγους όμως από τον συνάδελφο Μίντελμπουργκ, εμείς όπως ξέρετε είμαστε κατά των μακροοικονομικών προϋποθέσεων ε, και όπως είπε και η συνάδελφος Κωνσταντσα Κρέλ αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο εμείς, ε, με το οποίο δεν συμφωνούμε στην νέα πρόταση, όμως ε, για να το πω απλά θα μπορούσαν να ήταν χειρότερα τα πράγματα. Με βάση τις προκλήσεις που υπάρχουν, το Brexit, ε, τις περικοπές, τα το θέματα του περιβάλλοντος, της ένταξη, τη κοινωνική κοινωνικής πρόκειται για μια καλή πρόταση. Πρόκειται για μια καλή βάση συζήτησης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα εδώ στην, επιστροφή, στην, Επιτροπή Ρέτζη. Να ξεκινήσω με τα θετικά σημεία λοιπόν. Εμείς εδώ και πολύ καιρό δίνουμε μάχη για αυτά που υπάρχουν στην πρόταση αυτή τη στιγμή. Καταρχήν η ενίσχυση ε, της ε, Χρηματοδότηση ε, για τον στόχο 25% σχετικά με, τα, με την κλιματική αλλαγή. Θα μπορούσαν περισσότερα βέβαια. Εμείς ζητήσαμε περισσότερα, αλλά είναι ένα καλό βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης το γεγονός ότι τώρα θα έχουμε έναν καλύτερο ε, και έναν μακρύτερο αρνητικό κατάλογο. Δηλαδή τι δεν πρέπει να ξοδεύουμε στα πλαίσια των Ταμείων Συνοχής. Πριν είχαμε ένα μικρό κατάλογο, τώρα έχουμε όμως ένα μεγαλύτερο ε, σε ό,τι αφορά τις κακές επενδύσεις, ε, δηλαδή ορυκτά καύσιμα, αεροδρόμια, ε, χωματερές κτλ. Ο νέος, η νέα κλίδα κατανομής και η διεύρυνσή της είναι κάτι που εκτιμούμε ιδιαίτερα. Δώσαμε μάχη γι' αυτό. Δηλαδή να πάμε πέρα από το ΑΕΠ, να μην χρησιμοποιούμε ως μοναδικό κριτήριο δηλαδή το ΑΕΠ το κατακεφαλήν ΑΕΠ για την κατανομή των κονδυλίων, να λάβουμε υπόψη μας ε, την ενεργεία των νέων, την εκπαίδευση, τις κλιματικές συνθήκες, τα μέτρα ένταξης. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά θετικά για την ποιότητα των δαπανών ε, των Ταμείων συνοχή και βεβαίως το γεγονός ότι όλες οι περιφέρειες είναι επιλέξιμες και αυτό το είπαν και άλλοι. Επίσης χαιρόμαστε διότι η αρχή της εταιρική σχέσης, της σύμπραξη ε, επανέρχεται στην πρόταση διότι εμείς ως πράσινοι ε, είχαμε ανησυχήσει μετά την διαρροή που υπήρξε την περασμένη εβδομάδα όπου αυτή η υποχρέωση που υπήρχε ε, να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνία των πολιτών, οι τοπικοί και οι περιφερειακοί φορείς ε, και αρχές ε, σε κάθε βήμα από τον προγραμματισμό στην εφαρμογή δηλαδή των προγραμμάτων, κάτι που για μας ε, ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα, θετικό βήμα σε αυτήν την περίοδο. Δεν υπήρχε στην εκδοχή που είχε διαρρεύσει, σας στείλαμε άμεσα μια επιστολή, αλλά και σε άλλους συναδέλφους στην Κομισιόν. Χαιρόμαστε λοιπόν ιδιαίτερος που αυτή η αρχή επανήλθε στο κείμενο. Από την άλλη όμως μας λείπει κάτι άλλο, ε, κάτι εξαιρετικά σημαντικό, οι οριζόντιες αρχές στα άρθρα. Οι οριζόντιες αρχές όπως η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, η μη διάκριση, η βιώσιμη ανάπτυξη, αυτά δεν υπάρχουν πλέον στο διατακτικό του κειμένου ε, σε ένα άρθρο είναι κατακρεματισμένο σε διάφορα σημεία της πρότασης, ε, στην επιλογή των project, αλλά μόνο μερικός. Και αυτό αποτελεί αποδυνάμωση των οριζόντιων αρχών μας. Και αυτό είναι και το πρώτο μου ερώτημα, κυρία Επίτροπε. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι αυτές οι οριζόντιες αρχές, ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, μη διάκριση, βιώσιμη ανάπτυξη, ε, δεν θα αποδυναμωθούν εφόσον δεν υπάρχουν σε ένα άρθρο, αλλά υπάρχουν μόνο σε εκτιμώντας του κειμένου και ποιος είναι ο λόγος για την διαγραφή αυτών των οριζόντιων αρχών στο διατακτικό του κειμένου. Ε, είναι για λόγους απλοποίησης. Ε, δεν είναι μόνο απλοποίηση αυτό όμως, είναι αλλαγή πολιτικής. Είναι αποδυνάμωση μιας πολύ σημαντικής πολιτικής για μας. Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό και πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι αυτές οι οριζόντιες αρχές θα εφαρμοστούν. Και το δεύτερο ερώτημά μου, πάλι σύντομα, ε, διότι δεν έχει σχέση με, την CPR, με το CPR, έχει σχέση με τα, με τα ταμεία συνοχής. Είπατε στη συνέντευξη τύπου στις, ε, ότι στι 6 Ιουνίου η πρόταση Invest EU, το Ταμείο Αυτό Επενδύσεων, ε, είτε ενσωματωθεί εκεί το Ταμείο Juncker είτε όχι, θα παρουσιαστεί λοιπόν στις 6 Ιουνίου. Ξέρετε, έχει, δώσει μια μεγάλη, έχει δοθεί μια μεγάλη μάχη έτσι ώστε στον κανονισμό Omnibus να μην υπάρχει αυτή η αναλλακτική δυνατότητα να μεταφέρονται χρήματα από τα ταμεία συνοχή προ το ταμείο Juncker. Μπορείτε να μα εξασφαλίσετε ότι αυτή η δυνατότητα, το είπε ο κ. Κατάινεν στη συνέντευξη τύπου, αυτή η δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίων θα περιοριστεί αυστηρά και θα είναι αυστηρός εθελοντική για τα κράτη-μέλη. Ούτε με αυτό συμφωνούμε ακριβώς, αλλά είναι κρίσιμη σημασίας ε, για μας. Παρακαλώ να μας το εξηγήσετε, διότι είναι μια σημαντική, σημαντική παράμετρο στην όλη αυτή η συζήτηση της πολιτικής συνοχής για μας τους ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μόνικα για τα πλήρη αυτά σχόλια για την ΚΟΕ τώρα ο Δημήτρης Παπαδημούλης έχει το λόγο, παρακαλώ. Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι ε, προσωπικά εκτιμώ ιδιαίτερα την προσπάθεια της Επιτρόπου μέσα σε ένα πάρα πολύ ασφεκτικό πλαίσιο να βρει την καλύτερη δυνατή ισορροπία. Γιατί γνωρίζω καλά ότι και μέσα στην Κομισιόν υπάρχουν φανατικοί αντίπαλοι των πολιτικών συνοχής που προσπαθούν με κάθε ευκαιρία, και το Brexit είναι μία από αυτές, να περικόψουν τις πολιτικές συνοχές. Ξεκινώ από τα αρνητικά, κυρία Επίτροπε. Είμαι κατηγορηματικά αντίθετος και εγώ και η πολιτική μου ομάδα, αλλά και η μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη μείωση των κονδυλίων στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τις πολιτικές συνοχές. Πιστεύουμε ότι είναι λάθος η περικοπή των πολιτικών συνοχής. Και νομίζω ότι αν θέλουμε να αποφύγουμε μια παγίδα που μας έχουν στήσει, να αρχίσουν να τσακώνονται οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, τα νέα μέλη της διεύρυνσης για το πώς θα μοιράσουμε τη μειωμένη πίτα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι το Ευρωκοινοβούλιο να επιμείνει τους επόμενους μήνες στη θέση του ούτε ένα ευρώ μείωση της πολιτικής συνοχής. Αντίθετα, χρειάζεται ενίσχυση των πολιτικών συνοχή. Το δεύτερο αρνητικό είναι η αιμονή, όπως σημείωσε και η κυρία Κρέλ και η κυρία Βάνα, σε αυτή τη λογική της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας, η οποία είναι όχι απλώς αντίθετη με την θέση που επανειλημμένα το Ευρωκοινοβούλιο έχει υιοθετήσει, και φυσικά και η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, αλλά είναι αντίθετη και με την κοινή λογική. Είναι αντίθετη με τα διδάγματα που μας δίνει η εμπειρία. Σας θυμίζω ότι πριν τρία περίπου χρόνια η Κομισιόν ετοιμαζόταν να περικόψει τα κονδύλια των πολιτικών συνοχής για την Πορτογαλία και την Ισπανία με όπλο την περίφημη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Απέφυγε να το κάνει και το γεγονός ότι ήταν λάθος η περικοπή αποδείχθηκε από την εξέλιξη, από το πώς πάνε τα πράγματα στην οικονομία και στις πολιτικές συνοχές και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία και στη χώρα μου την Ελλάδα όπου η εφαρμογή κάποιων εξαιρετικών ρυθμίσεων έχει φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα και η Ελλάδα είναι σήμερα πρώτη σε ρυθμούς απορρόφησης και παραγωγικής αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων χάρη στο ότι εφαρμόστηκε με ένα ανοιχτό μυαλό και όχι με δογματικό τρόπο η πολιτική συνοχής. Άρα πρέπει να δούμε με βάση την κοινή λογική ότι χρειάζεται αυτά τα πράγματα περισσότερη ευελιξία. Έρχομαι τώρα σε κάποια πράγματα που τα θεωρώ θετικά. Νομίζω ότι είναι θετική η αλλαγή στην κλίδα κατανομής του λεγόμενου συστήματος του Βερολίνου. Είναι σωστό και υπόθηκε και από άλλους συναδέλφους άλλων πολιτικών ομάδων ότι εκτός από το ΑΕΠ μπαίνουν και άλλα κριτήρια. Οι χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανεργία νέων, που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή, που έχουν μεγαλύτερα προβλήματα για την ένταξη των μεταναστών ή τη στήριξη των προσφύγων δικαιούνται μεγαλύτερη βοήθεια γιατί έχουν περισσότερες ανάγκες. Και αυτό είναι θετικό και πρέπει να το στηρίξουμε μακριά από μια λογική εθνικών εγωισμών. Όπως επίσης θεωρώ θετικό ότι γίνεται μια προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών, αλλά με διατήρηση και των αναγκαίων ελέγχων, έτσι ώστε να διασφαλίζουν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι κυβερνήσεις και οι περιφέρειες ότι τα χρήματα αυτά που δίνονται για τις πολιτικές συνοχής θα πιάνουν πραγματικά τόπο, θα πηγαίνουν στους πολίτες. Γιατί βλέπουμε και περιπτώσεις όπου καμιά φορά δεν γίνεται αυτό και πηγαίνουν προς άλλες κατευθύνσεις. Έρχομαι, για να μην μακρηγορήσω, σε ορισμένες ειδικέ παρατηρήσεις. Νομίζω ότι για την τεχνική βοήθεια είναι ευπρόσδετα τα flat rates, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό να πάμε σε ένα ποσοστό πλαφών 2,5%. Νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνει στο 4%, γιατί έχουμε πολλά κράτη-μέλη που χρειάζονται τεχνική βοήθεια, καινούρια κράτη-μέλη, για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν παραγωγικά τους πόρους. Άρα να μείνει το 4% γιατί το 2,5% παραπέμπει σε ιδανικές συνθήκες διοίκησης που δυστυχώς δεν ισχύουν. Το δεύτερο είναι ότι δεν συμφωνώ με την μετατροπή του κανόνα νήσιν 3 σε νήσιν 2. Η πραγματικότητα έχει δείξει ότι δεν οδηγεί αυτό σε ταχύτερη υλοποίηση. Γι' αυτό και υιοθετήσαμε τον ΙΣΙΝ 3. Επομένως, ας επιδιώξουμε την βελτίωση της πραγματικότητας στην ε, πραγματική ζωή, την βελτίωση των επιδόσεων και όχι να αλλάξουμε έναν κανόνα που έχουμε θεσπίσει επειδή ακριβώς η πραγματικότητα μας το επέβαλε. Επίσης, πιστεύω ότι ο γενικός κανονισμός πρέπει να αφορά και το Rural Development Fund. Η εξαίρεσή του μου φαίνεται προβληματική. Και τέλος, διαφωνώ κατηγορηματικά με τις περικοπές στο Ίντερεγ. Νομίζω ότι το Ίντερεγ χρειάζεται ενίσχυση και όχι περικοπές και αυτό είναι και αναγκαίο εργαλείο για να υπηρετήσουμε και ευρύτερους στόχους ευρωπαϊκής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, τη διεύρυνσή της προς τα Δυτικά Βαλκάνια αν δεν ενισχύσουμε τα προγράμματα Interreg, πώς θα υπηρετήσουμε το στόχο αυτής της πολιτικής. Σας ευχαριστώ. Merci Ευχαριστούμε. Κύριε Επίτροπε, είδατε ότι έχουμε πολλές ερωτήσεις, ε, οι οποίες είναι ακριβείς. Μεταφέρουν ανησυχίες των συναδέλφων. Και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο να απαντήσετε στο πρώτο αυτό γύρο ερωτήσεων και μετά θα δώσουμε τον λόγο σε άλλους ομιλητές για το δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ. Καταρχήν, σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις, παρατηρήσεις, ιδέες που πάντοτε είναι χρήσιμες. Γιατί είστε άνθρωποι που καταλαβαίνετε αυτή την πολιτική, γνωρίζετε τις δυσκολίες. Θα ξεκινήσω με αυτό που είπε η κυρία Βάνο, ότι θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα τα πράγματα. Επί ένα χρόνο προσπαθούμε να επιτύχουμε τα σωστά αποτελέσματα. Περάσαμε από διάφορες φάσεις. Προετοιμάσαμε 20-25 διαφορετικά σενάρια μέχρι να καταλήξουμε κάπου. Αυτό το οποίο σας παρουσιάζουμε τώρα είναι το πιο ρεαλιστικό και το πιο φιλόδοξο σχέδιο σε σχέση με όλες τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις. Και μην ξεχνάτε από εκεί που, καταλή... από εκεί που ξεκινήσαμε ένα χρόνο πριν. Θα ήταν τραγικό να κοπεί κατά το ίμιση η περιοχή η πολιτική συνοχής, γιατί ακούγονταν τέτοιε φήμες. Βέβαια δεν μπορούν να είναι όλοι ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα. αλλά η λύση την οποία σας προτείνουμε τώρα πραγματικά είναι η πιο ρεαλιστική και η πιο φιλόδοξη. Θέλαμε να κάνουμε τις κατάλληλες προσαρμογές για να αποφύγουμε μεγάλες απώλειες. Ξεκινήσαμε, παραδείγματο χάρη, με ένα σενάριο για να περάσουμε από το μείον 45 στο συν 45 να περιορίσουμε απώλειες και ωφέλη. Οι ερωτήσεις σας είχαν μεγάλη ακρίβεια και θα προσπαθήσω και στις απαντήσεις μου να είμαι ακριβής. Για την κατηγορία των περιφερειών που ρώτησε ο κ. Σόλμπριχ, Έχουμε τον ίδιο αριθμό επιλέξιμων χωρών για το Ταμείο Συνοχής. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες με ΑΕΠ κάτω από 75% δεν αλλάζουν. Έχουμε καλύτερη συγκέντρωση σε αυτή την προγραμματική περίοδο στις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Το 75% των 374 δισεκατομμυρίων πάει στις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. 125 εκατομμύρια πολίτες ζουν σε αυτές τις λιγότερο ανεπτυγμένες ε, περιοχές σήμερα. Θα μειωθεί ο πληθυσμός στο μέλλον, αλλά η μείωση πληθυσμού ε, δεν επηρεάζει τη μεγάλη συγκέντρωση χρημάτων σε αυτές τις ε, περιοχές. Δεν συμφωνώ λοιπόν με την παρατήρηση σας ότι αλλάζει η πολιτική συνοχή, ότι αλλάζει η κατεύθυνση της πολιτικής. Τις ίδιες γραμμές ακολουθούσαμε από την αρχή και στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους και τώρα. Αν είχαμε χρησιμοποιήσει τη φόρμουλα του Βερολίνου αυτή καθεαυτή, σας διαβεβαιώ ότι θα ήταν πολύ μεγαλύτερες οι απώλειες από ό,τι αυτές που σας προτείνουμε. Γι' αυτό Είπαμε, χρησιμοποίησαμε αυτό που έχουμε συζητήσει και εδώ, ότι το κατακεφαλήνα ΕΠ δεν είναι ο μοναδικός παράγων και έχουμε και αυτούς τους δείκτες που θεωρούμε ουσιαστικούς για κάθε περιφέρεια, για την εκπαίδευση, για την ανεργία, για την κλιματική αλλαγή, για τη μετανάστευση γιατί αυτά όλα είναι ε, κίνητρα για τον πληθυσμό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου έχουμε τόσο μεγάλες αλλαγές στις περιφέρειες. Στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη, έχουμε περιοχές όπου έχει διπλασιαστεί ο πληθυσμός. Αν δείτε λοιπόν μηδέν στα χαρτιά, στην πραγματικότητα δεν είναι μηδέν, γιατί έχει διπλασιαστεί ο πληθυσμός και κάποιες περιφέρειες μπορεί να χάνουν σχεδόν 50%. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους. Όσον αφορά τις περικοπές, συμφωνώ μαζί σας. Οι περικοπές στην πολιτική συνοχή είναι μείον 10 σε πραγματικούς όρους. Αλλά υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού με το Brexit, χωρίς το Brexit, σε διαρκείς τιμές, σε τρέχουσες τιμές, με πληθωρισμό, χωρίς πληθωρισμό οι συνολικές περικοπές γενικά είναι μείον 10% όπως το υπολογίζουμε εμείς. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να εστιάζουμε τους πόρους ε, στα, ε, στα περισσότερο φτωχά κράτη-μέλη και περιοχές και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Η κατανομή πόρων αντανακλά τις ανισότητες ε, και την εξέλιξή τους. Αυτή είναι η λογική της πολιτικής συνοχής. Στα κράτη-μέλη και περιφέρειες όπου υπάρχει πρόοδος, μειώνεται σταδιακά η υποστήριξη της πολιτικής συνοχής και αντιστρόφως όπου έχουν επιδεινωθεί οι συνέπειες, αυξάνεται κάπως η στήριξη. Για το Ταμείο Συνοχής, άλλη μια ερώτηση του κυρίου Όλμπριχ σχετικά με αυτό, το Ταμείο Συνοχής δίνει σημαντικούς πόρους για τις αναπτυξιακές ανάγκες κρατών μελών στον τομέα του περιβάλλοντος και των υποδομών. Ξέρετε πολύ καλά ότι το Ταμείο Συνοχής σχεδιάστηκε για τα κράτη-μέλη που μπήκαν το 2004 όπου οι ανάγκες υποδομών για επεξεργασία αποβλήτων, για ε, σιδηροδρομικές μεταφορές, ε, για σιδηροδρομικές συνδέσεις, ε, υπήρχαν μεγάλες ανάγκες και τις αναπτυξιακές αυτές ανάγκες τις παρακολουθεί το Ταμείο Συνοχής και προσαρμόζεται. Ήταν ε, πολύ ε, εποφελής οι επενδύσεις και τώρα σε αυτά τα κρατημέλη όπως περιοχές ε, στην Πολωνία, Ουγγαρία κλπ. Όλες τις χώρες που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 προσαρμόζονται ε, οι πόροι και λαμβάνουν υπόψη ανάγκες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από τα δοτικότητα της ενέργειας, ε, παιδεία κλπ. Επιστρέφουμε στην κανονική κατανομή όπως προκύπτει από τη μέθοδο αλλά σε μεταξύ ε, αυξάνονται οι πόροι από το Περιφερειακό Ταμείο και το Κοινωνικό Ταμείο. Μπορεί να υπάρχουν λιγότερες ανάγκες υποδομές ε, και περιβάλλοντος στις χώρες αυτές. Μειώνεται λοιπόν η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής, αυξάνεται το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Κοινωνικό Ταμείο. Κωνσταντς, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κέλ για τα σχόλια που έκανε. Για την μακροοικονομική αιρεσιμότητα αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Κοινοβούλιο έχει διαφορετικές απόψεις ε, επί του θέματος. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε αυτό το μέτρο για να προωθήσουμε ε, την ε, ορθή διακυβέρνηση. Δώσατε το παράδειγμα της Ιταλίας. Δεν ξέρω αν η Ιταλία θα είχε ετοιμάσει ε, τον οδικό χάρτη για την υγεία. Ε, η Ιταλία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν το λέω μόνο για την Ιταλία. Αλλά αυτή η μακροοικονομική αιρεσιμότητα έχει λειτουργήσει ως σημαντικό εργαλείο για να διασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις μας πιάνουν τόπο. Ήδη στην περίοδο 2014-2020 έχουν επιτευχθεί πολλά στο πλαίσιο της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας και οι κυρώσεις ε, είναι αντίστοιχες των δεσμεύσεων. Εμείς ως Επιτροπή έχουμε το καθήκον να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την ορθή χρήση. Πολύ συχνά τα αποτρεπτικά μέτρα υπάρχουν για να μην χρησιμοποιούνται ποτέ. Κατανοώ τα ερωτήματά σας, αλλά εμείς ως Επιτροπή έχουμε το καθήκον να διασφαλίζουμε ότι τα χρήματα τα οποία επενδύουμε θα πρέπει να μεγιστοποιούν τον αντίκτυπο των επενδύσεών μας. Όσον αφορά το συνολικό προϋπολογισμό, έχει μειωθεί κάπως. Και όσον, ε, ε, ε, όσον αφορά την διασυνοριακή συνεργασία, έχουμε απλουστεύσει τις διαδικασίες. Τώρα όλες οι περιφέρειες μπορούν να συνεργάζονται και για τις πέντε προτεραιότητες με άλλες περιφέρειες με τις οποίες επιθυμούν να συνεργάζονται σε οποιαδήποτε περιοχή της Ευρώπης. Δεν μειώσαμε λοιπόν τη διασυνοριακή συνεργασία, αλλά αυτή η εδαφική συνεργασία είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε να την υποστηρίζουμε. Για το αποθεματικό απόδοσης, Θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω στην περίοδο μετά του 2020. Στην ενδιάμεση αναθεώρηση δεν θα ασχοληθούμε μόνο με το 6% αλλά και με όλες τις άλλες δεσμεύσεις, τις υποχρεώσεις μέχρι το 2026-2027. Ε, ξέρετε ότι το αποθεματικό απόδοσης ε, ήταν αρχικά ε, αυτόματο και δεν χρειαζόταν να λάβει υπόψη τις ειδικές συστάσεις αναχώρα ούτε το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο. Και αυτή η ακαμψία του συστήματος έπρεπε να αρθεί. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το νέο σύστημα δίνει ισχυρά κίνητρα ενώ παράλληλα τονίζει τις στρατηγικές κατευθύνσεις του αποθεματικού απόδοσης. Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της απόδοσης και για την υποβολή εκθέσεων, στην επόμενη προγραμματική περίοδο, το πλαίσιο απόδοσης θα καλύπτει όλα τα αποτελέσματα και τους δείκτες των προγραμμάτων. Όπως σας είπα, πολλές φορές στα κράτη-μέλη που επισκέπτομαι, λυπάμαι διότι βλέπω μερικές φορές ε, ότι αποτρέπονται από τη χρήση των κονδυλίων λόγω των ε, διαδικασιών ελέγχου και από την Επιτροπή και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Υπάρχουν λοιπόν και διάμεση ε, στόχοι, ορόσημα τέλος του 2024 και θα ληφθούν υπόψη τα επιτεύγματα κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση των προγραμμάτων το αποθεματικό ε, ε, απόδοση θα σταματήσει μετά το 2020 και στην ενδιάμεση αναθεώρηση θα εξετάσουμε ε, την περίοδο εφαρμογής και την ευελιξία και πώς μπορούμε να επανεξετάσουμε την ευελιξία του προγράμματος και θα αναλάβουμε υπόψη νέες προκλήσεις ούτως ώστε να προγραμματίσουμε την κατανομή μέχρι το 2027. Θα συνεχίσουμε να έχουμε μηδενική ανοχή στην απάτη. Αυτό ε, είναι αναμφισβήτητο. αλλά θέλουμε το πρόγραμμά μας να είναι φιλικό προς τους χρήστες και θέλουμε να έχουμε αυτό τον ε, ενιαίο έλεγχο για να, έχουμε, για να προωθήσουμε ε, την παρακολούθηση των επιδόσεων ώστε να έχουμε ε, αξιόπιστους δικαιούχους των προγραμμάτων μας. Μιλάμε για μεγάλα χρηματικά κονδύλια, επομένω προφανώ θα έχουμε μηδενική ανοχή στην απάτη. Για την ε, οριζόντια αρχή, επανέρχομαι στην κυρία Βάνα, η ισότητα των φύλων είναι πολύ σημαντικό, οι μη διακριτικέ μεταχειρήσει, οι εταιρικέ σχέσει, οι οριζόντιε αρχέ όπω η ισότητα των φύλων και η μη διακριτική μεταχείριση ε, εμφανίζονται πολύ περισσότερο στο νέο νομοθετικό πακέτο. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχει σημασία αν το αναφέρουμε ή όχι. Αυτή η αρχή πρέπει να τηρείται ούτως ή άλλως. Είναι κομμάτι του κοινοτικού κεκτημένου. Υπάρχει ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα έχουμε λοιπόν υποπαρακολούθηση το κατά πόσο τηρούνται αυτές οι αρχές, αναφέρονται εξ αρχής αλλά είναι δεσμευτικό να τηρούνται από τις αρχές υλοποίησης των προγραμμάτων. Ξέρετε ότι στην εταιρική σχέση υπάρχει αυτή η αρχή για την ισότητα των φύλων και για τη μη διακριτική μεταχείριση και πρέπει να τηρείται και στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση και στις ε, ε, συνθήκες εφαρμογής είναι ο καλύτερος τρόπος για να λειτουργήσει στην πράξη αυτή η αρχή. Δεν είναι συμβολική αρχή. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πολύ σημαντικές αρχές και πρέπει και στην πράξη να τηρούνται. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αν μένουν άλλα θέματα για τις προτεραιότητες, κυρία Βάνα. Το μεγαλύτερο τμήμα των κονδυλίων από τα 374 εκατομμύρια ε, ε, ευρώ θα πάει στις προτεραιότητες για την ευφυή Ευρώπη, καινοτομία και έρευνα και το δεύτερο για μια πιο πράσινη Ευρώπη για την ενέργεια, αποδοτικότητα ενέργειας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και για το EU Invest, ο Αντιπρόεδρος Κατάινεν Ε, αναφέρθηκε σε αυτό, θα υπάρχει μια ε, εθελοντική συμμετοχή και υπάρχει το όριο του 5%. Μπορεί να χρησιμοποιείτε το 5% του ΕΤΠΑ για το InvestEU. Προς τον κύριο Παπαδημούλη. Κανείς δεν συμφωνεί με τις μειώσεις, όντως, ε, αλλά τι να κάνουμε, και με την περίπτωση της Ελλάδας ξέρετε πολύ καλά ότι λάβαμε αυτά τα έκτακτα μέτρα και η Ελλάδα μπορεί τώρα να είναι υπερήφανη για την απορρόφηση κονδυλίων στην περίοδο 2014-2020 χάρη στη δουλειά της Επιτροπής Ρέτζη και χάρη στο Συμβούλιο και χάρη στην Επιτροπή έχει την υψηλότερη αποδοτικότητα, την υψηλότερη απορρόφηση στα έτη 2014-2020 και για την Ελλάδα και για την Ισπανία και για την Πορτογαλία. Η εμπειρία μας δείχνει ότι πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Υπάρχουν και έκτακτες περιστάσεις και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε γρήγορα. και κάποιες ε, ε, υποθέσεις ε, στη Γαλλία μας έδειξαν ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δείξουμε ευελιξία, όπως είδαμε στην περίπτωση Κατεπίλα. Τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ χειρότερα αν δεν είχαμε κάνει τις προσαρμογές και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι πρέπει να έχουμε κάποιους δείκτες. Ακόμη και σε πλούσιες χώρες έχουμε θύλακες φτώχες και χαμηλά ποσοστά εκπαίδευσης. Έχουμε βάλει λοιπόν 80% κατά κεφαλήνα ΕΠ και έχουμε ποσοστό ε, εκπαίδευσης, κλιματική αλλαγή ε, ε, ανεργία. Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τις τεράστιες ε, απώλειες και τα τεράστια ωφέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις τόσο ακριβείς και ε, απαντήσεις που απευθύνθηκαν μάλιστα και προσωπικά σε όλους τους ομιλητές. Ε, έχουμε περιορισμένο χρόνο διότι 15 ακόμα συνάδελφοι ζητούν το λόγο. Θα σας ζητήσω λοιπόν, αν θέλετε η Επίτροπος να προλάβει να σας απαντήσει, να είστε περιληπτικοί με σύντομες παρεμβάσεις κάτω το δυνατόν. Ιδανικά ένα με 1,5 λεπτό αναομιλτή. Ο λόγος στο συνάδελφο Φερνάντες, Επιτροπής Προπολογισμών. Ευχαριστώ πολύ ε, την Επίτροπο η ερώτησή μου είναι λίγο προκλητική. Ε, θα διατηρήσετε το πολιτικά το, το, το όνομα της συνοχής, γιατί αυτή η πολιτική δεν είναι πολιτική συνοχής. Η μείωση κατά 45% των πόρων του Ταμείου Συνοχής είναι καταστροφή της πολιτικής αυτής. Η πολιτική αυτή είναι για τους πιο φτωχούς. Και εσείς λέτε ότι πάει καλά. Αν πάει καλά, γιατί τη μειώνουμε κατά 45%. Αν διατηρήσετε το επίπεδο του Ταμείου συνοχή και εφαρμόσετε τα ίδια κριτήρια, τότε το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ διαφορετικό. Εγώ θα μιλήσω εκ μέρους της χώρα μου. Διότι και εσείς δημοσιεύετε τα εθνικά ποσά και αν το κάνετε αυτό διατρέχουμε τον κίνδυνο να δηλητηριάσουμε τη συζήτηση. Γιατί καθένα από εμά θα εξετάσει το ποσό που αφορά τη χώρα του. Αυτό όμως που θα έπρεπε καταρχήν να συζητήσουμε θα έπρεπε να είναι οι αρχές και οι στόχοι. Το Λουξεμβούργο για παράδειγμα, η Αυστρία, οι κάτω χώρες, το Βέλγιο, η Δανία. Είναι φτωχές χώρες δεν βλέπουν καμία μείωση, μηδενική μείωση. Και λέω τα, τις χώρες διότι με υποχρεώνεται. Η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Εστονία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Λετωνία, η Πορτογαλία. Είναι ε, πλούσιες χώρες <laughs> γιατί βλέπουν τα ποσά να μειώνονται από 7 μέχρι 24%. Πού βρίσκεται η αναλογικότητα υφίσταται ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Όταν περικόπτουμε ένα σημαντικό ταμείο που αφορά τους πιο φτωχούς κατά 45% ό,τι και να κάνετε με τα υπόλοιπα το, τελικό αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα βέβαια τα πράγματα και αν ο κόσμος καταστρεφόταν αύριο θα ήμασταν ακόμα χειρότερα. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Ευχαριστώ. Θέλω να σας συγχαρώ και να σας παρουσιάσω ορισμένες σκέψεις μου. Επιπλέον αυτών που ήδη αναφέρθηκαν. Καταρχήν να αναφερθώ στα θετικά σημεία της πρότασης. Η θεματική συγκέντρωση των στόχων, η απλοποίηση των διαδικασιών, η μεγαλύτερη ευελιξία που φέρνει η πρόταση. Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι αλλού σε άλλους τομείς δράσης της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνονται σημαντικές αυξήσεις με την ίδια ρεσιμότητα, μακροοικονομική ρεσιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν πολιτικές αποφάσεις τελικά στην πολιτική συνοχή. Ε, διευκρινίστε μου το εξής. Διαφωνώ με τις μειώσεις με τις περικοπές. Γιατί η πολιτική συνοχής είναι πολιτική καταπολέμησης στόχιας, σύγκλησης κλπ. Ως Πορτογάλος λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω πώς θα τα εξηγήσω όλα αυτά εγώ στους εκλογές μου, στους μου στη χώρα μου. Μια πολιτική η οποία εδώ και δεκαετίες, την οποία εδώ και δεκαετίες προσπαθούμε να προασπίσουμε, δέχεται ένα σημαντικό πλήγμα. Πορτογαλία είναι μια χώρα σχετικά φτωχή. Εγώ μάλιστα προέρχομαι και από μια περιοχή ακόμα πιο φτωχή της Πορτογαλίας. Πώς μπορώ να δικαιολογήσω μια μείωση ποσών που λαμβάνουμε, ενώ άλλες χώρες και άλλες περιοχές πιο πλούσιες από εμά θα δουν τα κονδύλια τους να αυξάνονται. Ευχαριστώ. Κύριε Ζουλό. Ευχαριστώ Επίτροπε, για την παρουσίασή σας. Θα είμαι σύντομος, διότι έχουν τεθεί πολλές ερωτήσεις ήδη. Όλες οι προτάσεις που, οι προτάσεις που έγιναν εδώ και μερικές μέρες προφανώς δεν είναι τέλειες. Θα πρέπει να δώσουν περισσότερο χρόνο στον εαυτό μας να τις αναλύσουμε. Νομίζω όμως ότι η Κομισιόν έκανε κάποιες ε, γενναίες προτάσεις. Πολλές από αυτές μάλιστα ε, έχουν κάνει δεκτές ε, τις δικές μας, ε, τα δικά μας σχόλια σε εκθέσεις μας, παλιότερες εκθέσεις μας. Η διεύρυνση της κατηγορίας των περιφερειών που βρίσκονται σε μετάβαση είναι σημαντική. Είναι μια καινούρια αρχιτεκτονική που πιστεύω θα επιτρέψει να καλύψουμε καλύτερα περιοχές σε στασιμότητα κινδυνεύουν να μείνουν πίσω. Το ανέφερε αυτό και η 7η έκθεση συνοχής. Ένα άλλο θέμα όμως που θέλω να θίξω, εν συντομία, είναι το εξής. Πολλές περιοχές περιφέρειας Ευρώπης θα επηρεαστούν πολύ από το Brexit. Για παράδειγμα στην Ιρλανδία, αλλά και η Βρετανία, η Νορμανδία, η Haute France στη Γαλλία. Θα μπορούσατε να ε, θα μπορούσαμε να ε, διαθέτουμε κάποιο ιδιαίτερο εργαλείο για αυτές τις περιοχές στο μέλλον. Ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ μην ξεπερνάτε το χρόνο σας για να μπορούν να πάρουν το λόγο όλοι. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να κλείσουμε τον κατάλογο των μιλητών. Ο συνάδελφος Βόγκλ. Yeah, uh, um, όπως είπαν οι συνάδελφοι, το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ο προϋπολογισμός του, της πολιτικής συνοχής μετά το 2019. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα προσπαθήσει να αντιστρέψει ορισμένε από τι ε, περικοπέ που προτείνει η Κομισιόν. Ορισμένε ε, εθνικέ μειώσει είναι τεράστιε. Βέβαια, το Ηνωμένο Βασίλειο πλέον δεν θα είναι εδώ μετά το 2019, οπότε θα υπάρχει μείωση ε, των εσόδων ε, οπότε με αυτή την έννοια χρειάζεται να γίνουν κάποιες περικοπές. Τώρα, η Κομισιόν έχει κάνει πολύ καλές προτάσεις κατά τα άλλα και θα ληφθούν υπόψη στις διαπραγματεύσεις. Καλύπτονται για παράδειγμα όλες οι περιφέρειες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχουμε επιμείνει σε αυτό, ευελιξία και αυτό πολύ καλό. Και όσοι εισηγητή για την έκθεση των επιπτώσεων των, ε, των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην, στην Βόρεια Ιρλανδία θα ήθελα να συνεχιστούν να συνεχιστεί η χρηματοδότηση διότι βοηθάει την ερευνητική διαδικασία και η Κομισιόν και η Ιρλανδική κυβέρνηση τη στηρίζει αλλά και, το, και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αυτή τη χρηματοδότηση. Επίσης υποστηρίζουμε την απλοποίηση σήμερα και του μοναδικού, και του μοναδικού λογιστικού ελέγχου. Θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση πράγματι. Ένα μια τελική ερώτηση, τελευταία ερώτηση για το Interreg. Η πρόταση φαίνεται να εστιάζεται στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που έχουν χερσαία σύνορα. Αυτή είναι η πρόθεση του Ιντερεγ μόνο. Αυτό θα είναι, αυτή θα είναι η, η πρόθεση του Ιντερεγ στο μέλλον ή θα συμπεριληφθούν και χώρες που έχουν θαλάσσια σύνορα μεταξύ τους. Ευχαριστώ η Μαρτίνα Άντερσον έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ κυρία Επιτροπέ που είστε εδώ σήμερα. Θα ήθελα να αναγνωρίσω πραγματικά ε, και να συμφωνήσω με αυτό που είπατε στην συνέντευξη τύπου σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της ειρήνης στην Βόρεια Ιρλανδία. Ήμουν και στην αποστολή μεταξύ των Ευρωβουλευτών. Εκεί είδαμε τον αντίκτυπο της ε, πολιτικής συνοχής και της χρηματοδότησης της ειρηνευτικής διαδικασίας στην χώρα αυτή. Βεβαίως δυσκολίες υπάρχουν, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν πάει κάποια χρήματα από περιφερειακά ταμεία και στο βόρειο Μπέλφαστ. Ε, θέλω να σας βοηθ... ευχαριστήσω ιδιαίτερα που είπατε ότι θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση και μετά το Brexit ε, αυτών των προγραμμάτων, διότι αυτή η διαδικασία ειρήνευσης ε, είναι εξαιρετικά σημαντική. Ξέρετε, η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής ε, είναι καλό να την έχει ο καθένας και να την διαβάζει. Σας δώσω μάλιστα ένα αντίγραφο. Ε, υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες. Ε, στην αποστολή αυτή είδαμε τις ανησυχίες, διότι υπάρχει ο φόβος ότι το Brexit θα βάλει τέλος μια εικοσαετή διαδικασία ειρήνευσης. Πρέπει λοιπόν αυτό που κάνει το Κοινοβούλιο να ακουστεί, να ακουστεί και στον κόσμο, να καταλάβει ο κόσμος ότι θα υπάρχει κάποια προστασία και μετά το Brexit. Υπάρχει και αρχή της σύμπραξης και οι ριζόντιες αρχές και άλλα που ήθελα να πω για την μακροοικονομική ρεσιμότητα, αλλά δεν προλαβαίνω. Από τους πράσινους τώρα, παρακαλώ, επόμενος ομιλητής, ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ στη σημερινή συνεδρίαση, κύριε Επίτροπε, να μην χαθεί χρόνο, οπότε να μην επαναλάβω αυτά που είπαν ήδη οι συνάδελφοι. Ήθελα μόνο να εκφράσω την έκπληξή μου, διότι πριν από δύο μήνε ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ολομέλεια είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποτέ δεν πρόκειται να συμφωνήσει με περικοπέ στην πολιτική συνοχή. Και τώρα οι προτάσει σα πάνε προ την αντίθετη κατεύθυνση. λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να επιλύσει όλα τα νέα προβλήματα που έχουν προκύψει εις βάρος της πολιτικής συνοχής. Εάν θέλουμε νέες εργασίες, <clears throat> να ανοίγουμε νέους φακέλους, χρειαζόμαστε καινούρια κονδύλια. Δεν μπορούμε να πειράζουμε κονδύλια από αλλού, διότι τα προηγούμενα προβλήματα θα διωγκωθούν. Είναι περίεργο πιστεύω, που η μείωση της πολιτικής συνοχής και των σχετικών κονδυλίων αφορά κυρίως τις χώρες που βρίσκονται σε μεταβατική φάση. Δηλαδή αυτές οι χώρες ε, ουσιαστικά θα επιστρέψουν πίσω με τους φτωχούς. Έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν ότι οι χώρες που βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια περίοδο στασιμότητας παγώματος της οικονομίας. Υπήρχε μια ανάπτυξη που βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό και στην ενίσχυση. Θα πρέπει να γίνεται πολύ πιο προοδευτικά αυτή η μείωση. Λέγεται ότι μειώνεται ο συνολικός προπολογισμό. Εντάξει, αλλά να μοιραστεί ισότιμα. Ναι, οι συντονιστές εξέφρασαν τις πολιτικές θέσεις της κάθε πολιτικής ομάδας. Οπότε παρακαλώ να πηγαίνετε κατευθείαν στο ερώτημά σας προς την Επίτροπο όταν παίρνετε το λόγο. Ο κ. Μπόγκοβιτς έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είχατε δύσκολη δουλειά, κυρία Επίτροπε, και θέλω να επικεντρωθώ σε ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Δεν υπάρχει κάποιο κριτήριο για το θέμα της μετανάστευσης μεταξύ περιφερειών και από τις πιο φτωχές προς, προς τις πιο πλούσιες περιφέρειες. Δεν υπάρχει τέτοιο κριτήριο. Πολλές περιφέρειες έχουν χάσει τον πληθυσμό τους. Αυτό το κριτήριο λοιπόν το χρειαζόμαστε στο Ταμείο Συνοχής. Αναφερθήκατε στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ε, ε, Γεωργικής Ανάπτυξης, ναι, Ανάπτυξης της Υπέθρου, ε, δεν είναι σωστό αυτό. Η Υπέθρος θα αδειάσει τελείως έτσι. Θα βρεθούν όλες τις πόλεις και δεν θα μείνει κανείς στα χωριά. Ταυτόχρονα έχουμε πολύ μεγάλα ποστά μετανάστευσης ε, παγκοσμίως και αυτό δημιουργεί πολλά ζητήματα, τα οποία προσπαθούμε εμείς να τα επιλύσουμε στη δική μου, στις δικές μας περιφέρειες και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην τελική πρόταση. Ευχαριστώ εν συντομία, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Επίτροπο. Το αποτέλεσμα αυτό δεν μας ικανοποιεί βεβαίως απολύτως, αλλά είναι γενικά θετικό. Διότι, και αυτό διότι εσείς δώσετε μάχη, μεγάλη μάχη. Έχω δύο ερωτήματα. Οι νέες κατηγορίες που αφορούν κριτήρια όπως η ανεργία, αυτές οι νέες παράμετροι, όπως περιπτώσει, λαμβάνονται υπόψη και στις τρεις κατηγορίες περιφερειών. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει να εγκριθεί το CFP και ο κανονισμός για τη συνοχή κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας σε πρώτη ανάγνωση τουλάχιστον διότι το χρονοδιάγραμμα έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις περιφέρειες. Κάτι ακόμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, εντάξει δεν έχουμε ακόμα τον κανονισμό, Έχουμε όμως την εντύπωση ότι πάμε προς μια επανεθνικοποίηση για τις περιφέρειες, η συνοχή και το κοινωνικό ταμείο είναι αλληλένδετα, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλος ο κίνδυνος εδώ. Τέλος, το ψήφισμα για τις περιοχές της Υπέθρου, τις ορεινές περιοχές, ε, θα εγκριθεί τον Ιούλιο. Μιλάμε για 80% του εδάφους της Ένωσης. Όμως οι πόλεις αντιπροσωπεύουν 80% του πληθυσμού. Τα εδάφια έχουν και αυτά τη σημασία τους. Πέρα από τις πόλεις ε, και τις αστικές περιοχές θα υπάρξει ένα πρόγραμμα για την Ήπεθρο, για τις ορεινές περιοχές, θα υπάρξει μια προσαρμογή των προτεραιοτήτων για να μπορούν ε, και οι αυτές οι περιφέρειες να χαίρουν προτεραιότητες. Ευχαριστώ ε, κύριε Μπάλετιτς, παρακαλώ, κυρία Μπάλετιτς, παρακαλώ σύντομα. Ευχαριστώ. Έχω πολλά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τον εφαρμοστικό κανονισμό, αλλά δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό. νη συνδύωση, χρηματοδότηση, προχρηματοδότηση, ερεσιμότητα, όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν. Να πω ότι ως Επιτροπή Ρέτζη αλλά και εσείς ως Επίτροπος δεν μπορείτε να είστε ικανοποιημένοι με αυτήν τη μείωση της πολιτικής συνοχής. Όταν εξετάζουμε το σύνολο του πολιτικού δημοσιονομικού προγράμματος βλέπουμε ότι έχουμε αύξηση στα προγράμματα ανταγωνιστικότητας. Και οι πιο αναπτυγμένες χώρες βεβαίως είναι αυτές που χρησιμοποιούν περισσότερο αυτά τα προγράμματα ανταγωνιστικότητας ε, ε, για προφανείς λόγους. Με τις περικοπές λοιπόν στην πολιτική συνοχή και με την αύξηση των προγραμμάτων ανταγωνιστικότητας στέλνουμε ένα εντελώ λανθασμένο μήνυμα. Δεν γίνεται δηλαδή ουσιαστικά εδώ δουλειά ε, ε των ανισοτήτων αλλά αύξησή τους. Δεν δρούμε αλληλέγγυα. Και κάτι ακόμα για αυτόν τον πίνακα κατανομής αναχώρα. Νομίζω ότι πραγματικά χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη φόρμουλα με στοιχεία για την κάθε χώρα για να καταλάβουμε καλύτερα πώς φτάνουμε σε αυτά τα ποσά για την κάθε χώρα. Διότι όταν βλέπω το επίπεδο ανάπτυξης, βεβαίω είπατε ότι λάβατε υπόψη σας και άλλους δείκτες, αλλά παρόλα αυτά ε, δεν μπορώ να βγάλω εγώ, να καταλάβω πώς φτάνει στο αποτέλεσμα αυτό. Ευχαριστούμε. Ζωζεφ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, λυπάμαι ιδιαίτερα για τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται αυτός ο διάλογος με την Επίτροπο. Είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο του προϋπολογισμού ε, να το λάβουμε υπόψη μας. Η Επίτροπος έχει έρθει να μας μιλήσει για το Ταμείο Συνοχής που αποτελεί το 30% του προϋπολογισμού. Και δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο και βιαζόμαστε για τη διεξαγωγή της συζήτησης. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, λυπάμαι. Θέλω να πω προς την Επίτροπο ότι γνωρίζω τη δέσμευσή σας και την αποφασιστικότητά σας υπέρ ε, των ε, συμφερόντων ε, των περιοχών και ιδίως των διαμερισμάτων, υπερπόντιων διαμερισμάτων και περιοχών της Γαλλίας. Υπάρχουν όμως δυνατότητες οι οποίες θα έπρεπε να προσφέρονται για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη των περιφερειών μας και από την πείρα μου θα σας πω ότι μία ε, δημοσιονομική πρόταση ε, στην πράξη είναι ε, η πολιτική βούληση. Όταν ξέρουμε τι περιμένει ο λαός, τι περιμένουν οι πολίτες και όταν αυτά τα οποία εμείς τους προσφέρουμε ε, υπολείπονται των προσδοκιών τους, υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει να έχετε τη βούληση και την αποφασιστικότητα να υποβάλλετε προτάσεις πολύ περισσότερο βελτιωμένες. Αυτά και για μας και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Ζωζεφ. Να υπενθυμίσω ότι αφιερώσαμε δύο ώρες στη συζήτηση με την Επίτροπο. Είναι λογικό να δίνουμε στους συντονιστές το χρόνο να εκφράζουν τη θέση των πολιτικών ομάδων και στην Επίτροπο το χρόνο να απαντήσει για τα όσα προτείνει η Επιτροπή θα δώσω το λόγο σε άλλους δύο ομιλητές. Η Επίτροπος δεν θα μπορέσει να απαντήσει με μεγάλη ακρίβεια σε όλες τις ερωτήσεις λόγω των, του χρονικού περιορισμού. Θα δώσουμε το λόγο όμως στην Επίτροπο να κάνει μια συνολική παρέμβαση στο τέλος και δίνω τώρα το λόγο στους επόμενους συναδέλφους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, καταρχήν προς την Επίτροπο θέλω να πω Ξέρω από πού ξεκινήσατε. Δεν ξεκινήσατε από το 0, αλλά από το μείον 10. Αυτό το οποίο επιτύχατε μπορεί να μην είναι τέλειο, αλλά είναι το καλύτερο δυνατό. Ξέρω ότι έχετε 4 λεπτά για να απαντήσετε σε 15 ερωτήσεις, άρα ε, θα πω το εξή. Εφόσον το κέντρο των αποφάσεων έχει μετακινηθεί στην οδό Βίρτ, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα που μιλάνε όλοι. Δηλαδή, πιστεύετε ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι ζουν σε μια περιοχή ΝΑΤΣ 2 που βρίσκεται σε μετάβαση, καταλαβαίνουν οι πολίτες ότι ζουν σε μια περιοχή που είναι επιλέξιμη για ένα πρόγραμμα διασυνοριακή συνεργασία. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα κανονισμό CPR που θα είναι εύκολο να διαβάζεται, σαν να διαβάζουν οι πολίτε εφημερίδα. Διαφορετικά, να μην αναρωτιόμαστε γιατί οι πολίτε πιστεύουν ότι η Ευρώπη είναι το μεγαλύτερο λάθο και μετακερδίζουν και εκλογέ όπω προσφάτω η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο είχαν δυόμιση χρόνια να εγκρίνουν το CVA την προηγούμενη φορά. Τώρα έχουμε οχτώ μήνε και ο χρόνο δουλεύει εναντίον μα, Άρα πρέπει κατευθείαν να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε. Αν κάπου υπάρχουν λιγότερα χρήματα θα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί είναι λιγότερα τα χρήματα. Μπορεί σε κάποιε περιφερειές να επενδύουμε εδώ και 20 χρόνια και να έχει καταλήξει σε καλά και θετικά αποτελέσματα. Θα πρέπει να εξηγούμε καλύτερα λοιπόν αυτά τα οποία κάνουμε διαφορετικά θα μιλάνε για τη φούσκα των Βρυξελών, για τη φούσκα του Στρασβούργου. Εμείς θα πρέπει να τη σπάσουμε αυτή τη φούσκα και πρακτικά να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι αυτό το CPR δεν είναι πάλι άλλο ένα χαρτομάνι, αλλά είναι κάτι που θα βελτιώσει τη ζωή τους τα επόμενα 7-10 χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφος Έτμαν. Αγαπητή κυρία Επιτροπέ, ε, η... αν ε, χρειάζεται την υποστήριξή μας για την καινούργια κλίδα κατανομής η Κομισιόν πρέπει να μας την εξηγήσει καλύτερα. Γιατί λέτε ότι στην ε, επόμενη προγραμματική περίοδο θα βοηθήσουμε τους πιο φτωχούς. Δεν βλέπω όμως τις, δεν καταλαβαίνω όμως τις προτάσεις. Δεν, ποιος θα καταλάβει ότι η Λιθουανία βλέπει τα κονδυλία της να μειώνεται κατά 25%, η Φιλανδία να αυξάνεται κατά 5%, ε, η Πορτογαλία να βλέπει μείωση και η Ισπανία να βλέπει αύξηση. Ε, πώς θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά στους πολίτες μας. Χρειαζόμαστε περισσότερες λεπτομέρειες, περισσότερες εξηγήσεις για, την καινούργια, ε, για την καινούργιο τύπο σύμφωνα με τον οποίο, ε, ε στον οποίο βασίζεται η κατανομή. Επίσης θέλουμε να μηδενίσουμε τις απάτες, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε και την ε, ε, ομαδική ε, ευθύνη, το συλλογική ευθύνη. Ευχαριστώ και Πλουσόφσκι. Κύριε Επίτροπε, έχω ένα τεχνικό αίτημα εξ ονόματος όλων πιθανώς. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, ερωτήσεις πολλές. Οπότε δεν θα θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα, παρόλο που έχω πολλά. Θέλω όμως να ζητήσω από τον Πρόεδρο και από εσά κύριε Επιτροπέ να ξανασυναντηθούμε την ερχόμενη εβδομάδα για να συνεχίσουμε τη συζήτηση γιατί όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά. Να σας υπενθυμίσω ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια επαναλαμβάνουμε μία και μοναδική δήλωση πόσο σημαντική είναι η συνοχή, πόσο σημαντικά είναι αυτή η πόρη και βλέπω, βλέπουμε να μειώνονται πολύ, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε. Δύο ώρες δεν είναι αρκετές. Ας ξανασυναντηθούμε την ερχόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Κλείνουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Είμαστε περιορισμένοι χρονικά, γνωρίζετε ότι θα πρέπει να πάμε στην Ολομέλεια γιατί ξεκινούν οι ψηφοφορίες σε λίγο. Σας δίνω το λόγο κυρία Επίτροπε για να απαντήσετε στα τελευταία σχόλια που έγιναν. Η Επιτροπός, καταλαβαίνω πολύ καλά το έτοιμά σας και πιστεύω πράγματι ότι πρέπει να σας εξηγήσουμε καλύτερα, να μιλήσουμε καλύτερα για αυτά τα πράγματα και εγώ και η ομάδα μου. Η Γενική Διεύθυνση, ο υπεύθυνο του προσωπικού μου γραφείου, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσει θέλετε να θέσετε. Γιατί πραγματικά πιστεύω θα πρέπει να μπορείτε να επιστρέψετε στις χώρες σας και να εξηγήσετε τους περιορισμούς που έχουμε, ε, τις προτεραιότητες, ε, την επίπτωση του Brexit και όλα αυτά. Τώρα, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δευτέρα και Τρίτη είμαι στο Τάλιν και την Πέμπτη στη Σόφια με τους υπουργούς για το Συμβούλιο. Αλλά θα μπορούσαν ενδεχομένω οι, οι συνεργάτες μας να βρουν την κατάλληλη στιγμή. Καταλαβαίνω όμως τις ανησυχίες σας. Πιστέψτε με ότι εδώ και μήνες προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία, ε, ψάχνουμε, αναζητούμε διάφορα σενάρια. Η, εξακολουθούμε να την ονομάζουμε πολιτική συνοχή πράγματι, γιατί είναι ε, η πεμπτουσία της αλληλεγγύης και αφορά όλες τις περιφέρειες. Το ζήτημα είναι να ισορροπήσουμε το κοινωνικό ταμείο, τα ταμεία συνοχής και το ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης. Όσο πιο πολλά δώσουμε στο Ταμείο Συνοχής, τόσο θα πρέπει να αφαιρέσουμε από τα άλλα δύο. Ε, για τις καινούριες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε κάνει ήδη πολλά πράγματα για υποδομές, ε, σιδηρόδρομο, οδικές ε, μεταφορές, δρόμους κλπ. Και αυτές οι χώρες χρειάζονται άλλου τύπου επενδύσεις πλέον. Οπότε γι' αυτό λόγο είπαμε ε, λιγότερο ταμείο συνοχής και περισσότερο ταμείο κοινωνικό ταμείο και ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης. Αν συμφωνήσουμε ότι η πολιτική συνοχή αφορά όλες τις περιφέρειες, τότε θα πρέπει να στηρίξουμε και την Αυστρία και τη Δανία, όπως είπατε. Και θα πρέπει να τους δώσουμε μια κρίσιμη μάζα. Οι κάτω χώρες παίρνουν 12 ευρώ ανακάτοικο. Πώς να τα μειώσουμε. Αν τους δώσουμε ένα μόνο ευρώ ανακάτοικο θα μας πούνε όχι ευχαριστώ. Σε άλλε χώρες το αντίστοιχο ποσό είναι 200 και 300 ευρώ ανακάτοικο. Οπότε χρειάζεται να διατηρήσουμε κάποιες ισορροπίες. Εφόσον αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε όλες τις περιφέρειες, πόσο να μειώσουμε τη Δανία και τις κάτω χώρες. Θα μας πούνε όχι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν το χρειαζόμαστε. Η... Στην ε, Δανία έχουμε 14 ευρώ ανακάτοικο, στις κάτω χώρες 12. Στις ε, χώρες συνοχής ε, το αντίστοιχο ποσό είναι 300 και 400 ευρώ ανακατοικο. Αυτή είναι η πολιτική συνοχή. Είναι πράγματι η έκφραση της αλληλεγγύης. Προφανώς δεν ήταν επιθυμία μας να επιβάλλουμε περικοπές. Προφανώς δεν μπορούμε να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα στην πολιτική συνοχή και δίνω μάχες με τους άλλους συναδέλφους στην Κομισιόν. Γιατί ο κάθε συνάδελφος θέλει να αφήσει μια κληρονομιά για το μέλλον, για την ιστεροφημία του, ε, πρικοδοτώντας με μεγαλύτερα ποσά το δικό του πρόγραμμα. Ψηφιακές οικονομίες, το ένα το άλλο. Ε, και δίνουμε μάχη για να διατηρήσουμε τα ποσά του Ταμείου Συνοχής, της Πολιτικής Συνοχής. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Σίγουρα ε, δεν είναι το ευκταίο με, με το πρόγραμμα για την ειρήνευση στην ε, Ιρλανδία, το Peace Plus. Λυπούμαστε που φεύγει το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά έδωσα μάχη για να διατηρηθεί αυτό το πρόγραμμα γιατί αποτελεί πολιτικό μήνυμα. Εμείς συνεισφέρουμε μεγάλο ποσό η Δημοκρατία της Ιρλανδίας συγκεκριμένα. Να δούμε τι θα βάλει και η άλλη πλευρά. Να δούμε πώς θα ανταποκριθεί το Ηνωμένο Βασίλειο στην επιθυμία μας, στην εκπεφρασμένη μας επιθυμία να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση. Για τη μέθοδο του Βερολίνου τώρα. Κυρία Μάλετιτς. Ε, σύμφωνα με την του Βερολίνου, ε, το ΑΕΠ, ε, κατά κεφάλι ΑΕΠ, σταθμίζεται με το, στο 80%. Αν θέλετε, κάντε μας μια επίσκεψη να σας δείξουμε ακριβώς τι κάναμε. Κάναμε μερικές διευθετήσεις, διότι αν είχαμε 100% ε, σταθμισμένο το ΑΕΠ, η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη. Τα ποσά της Πορτογαλίας θα μειωνόντουσαν κατά πάνω από 75%. Η μείωση αυτή τη στιγμή είναι 7%. Πολύ μικρότερη η περικοπή από το 10% που είναι η συνολική μέση μείωση. Η, τα ποσά των ταμείων μειώθηκαν ε, και λάβουμε υπόψη ε, θα λάβουμε μάλλον υπόψη τελικά ε, το πώς έχει προχωρήσει κάθε περιφέρεια. ορισμένες περιφέρειες στην ίδια χώρα θα πάρουν περισσότερα, άλλες λιγότερα. Μετά, το χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα είναι στα χέρια σας. Δεν είναι δικό μας δημιούργημα. Εμείς θέλουμε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία σε ένα χρόνο. Η σημερινή συζήτηση όμως δείχνει ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της πολιτικής συνοχής δεν είναι επαρκής για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Και γι' αυτό, αυτό το είναι εξ αρχής. Υπό αυτές τις συνθήκες πρέπει να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν περισσότερα, μεγαλύτερα ποσά για να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματα και τις ανάγκες των πολιτών μας. Αυτή τη στιγμή ο προπολογισμό έχει καταρτιστεί με βάση ε, το όριο του 1 ευρώ κατά και ανά ημέρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α πιέσουμε λοιπόν να, τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν μεγαλύτερα ποσά στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χρειαζόμαστε. Δεν μπορούμε ε, να κάνουμε τα πάντα με ένα ευρώ ανακάτοικο ένα ημέρα. Πρέπει να διευρύνουμε τους ιδίους πόρους μας. Στο Συμβούλιο όμως δεν συμφωνούν με το φόρο για την κλιματική αλλαγή. Αν δεν συμφωνούν λοιπόν με την αύξηση των ιδίων πόρων, θα χρειαστεί να αυξήσουν τη συνεισφορά τους. Για αυτή την προγραμματική περίοδο το 75% του προπολογισμού πηγαίνει στις λιγότερο αναπτυγμένε περιοχές, περιφέρειες. Κάτι που, είναι, που ε, αποτελεί αύξηση σε σχέση με την τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο. Λοιπόν, το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι το άριστο, αλλά είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρηθεί η πολιτική συνοχή ως πολιτική που θα αφορά όλες τις περιφέρειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να σας υπενθυμίσω ότι πρόκειται για μια πρόταση της Κομισιόν και είμαστε συνομοθέτες. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το Συμβούλιο. Οπότε αναλάβετε τις ευθύνες σας, του ρόλου σας ως συνομοθέτες και ας πιέσουμε τις, ε, τα κράτη-μέλη. Θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη 20 Ιουνίου στις 9 το πρωί. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλή ψηφοφορία και καλή επιστροφή στις χώρες σας.